Έτσι ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες για σήμερα. Τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περίοδου συνόδου.